Να προωθήσουμε λοιπόν τη συνεργασία με το Κοινοβούλιο, ιδιαίτερα με την Επιτροπή για την Ανάπτυξη του Κοινοβουλίου. Κομισιόν, τον κύριο Σεύκοβιτ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συζήτηση ολοκληρώθηκε. Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί αύριο το μεσημέρι στις 12. Καλή σας νύχτα.